Ο πρόεδρος ε, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Ρόσεν Πλεύνελιεφ. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε Λεβέινα, καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μεγάλη τιμή η παρουσία σας εδώ σήμερα. Για πολλά χρόνια ήσασταν σε στενή επαφή ως πρόεδρος της χώρας σας, που είναι σημαντικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλατε στις στενές σχέσεις. Και εδώ και δύο χρόνια αντιμετωπίζουμε από κοινού την πρόκληση της ε, μετανάστευσης. Σας ευχαριστώ πολύ για την επίσκεψή σας. Κύριε Πρόεδρε Πλευνέιεφ, είναι τιμή μας που είστε ε, εδώ στο Κοινοβούλιο. Έχετε το λόγο. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξοχότητες, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Είναι προνόμιο πραγματικά που βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα και απευθύνομαι σε εσά ως πρόεδρος της Βουλγαρίας.